και παρουσία της κυρίας Άστον όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έναντι της Κίνας, όσον αφορά αυτό το πρόβλημα, νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ ενδειγμένο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, κύριε Κονβέντιτ. Να το θέσετε αυτό, σας παρακαλώ, στη διάσκεψη των Προέδρων, ελεύθερα. Σαν Πρόεδρος της πολιτικής σας ομάδας έχετε αυτή τη δυνατότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θα προχωρήσουμε και θα πάμε στο πρώτο σημείο της σημερινής ημερήσιας διάταξης, η κοινή συζήτηση, Ευρω... η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 2009 και ισοτιμίες των διαφόρων νομισμάτων. Έχουμε την έκθεση BAU για την ετήσια BOLTS που είναι η ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του 2009 και έχουμε και δήλωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελευταίε εξελίξει διεθνεί συναλλαγματικέ ισοτιμίε. Ενωτήτω τη δηλώσεω τη Επιτροπή. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω ένα αίτημα να απευθύνω σε όλους σας. Εάν μας εγκαταλείπετε, σας παρακαλώ, αν μπορείτε να φύγετε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εγώ θα προτιμούσα να μείνετε μαζί μας, αλλά σας παρακαλώ, δώστε μας τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Το ταχύτερο δυνατόν παρακαλώ να αποχωρήσετε. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σας για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας, τη συζήτηση της Ολομέλειας. Συνάδελφε Κον Μπέντιτ, Ντάνιελ, σε παρακαλώ. It's very difficult to start. Okay. Our rapporteur. Ο εισηγητής μας ο συνάδελφός μας Μπουρκαρτ Μπάλτς. Έχετε το λόγο συνάδελφε. Ο κύριος Μπουρκαρτ Μπάλτς. Herr Präsident, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Κάποιοι είπε να κάνουμε λίγο ησυχία, ελπίζω να το τηρήσουν οι συνάδελφοι. Κυρίε και κύριοι, έχουμε σήμερα να συζητήσουμε την έκθεση κυρίω τη επιδόση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το 2009, κατά μια χρονική περίοδο δηλαδή κατά την οποία η χρηματοπιστωτική η οικονομική ε, κρίση ε, επηρεάζουν και τις ε, πολιτικές δράσεις βεβαίως. Η κρίση η οποία ήταν καθαρά χρηματοπιστωτική στην αρχή μετατράπηκε σε ένα δεύτερο κύμα, σε μια κρίση που έπληξε ολόκληρη την πραγματική οικονομία. Έχει περιοριστεί η οικονομική δραστηριότητα, πέφτουν ε, τα επιτόκια, ενισχύονται σημαντικά ε, τα ποστά χρέωση των ε, ιδιωτικών νοικοκυριών, η κατάσταση ιδιαίτερα της αυξημένης της υπερχρέωσης οδηγεί τις κυβερνήσεις σε σημαντικά πακέτα λιτότητας τα οποία ήταν απαραίτητα κατά την άποψή μου. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα θα έπρεπε από πολύ καιρό να είχαν ε, τεθεί σε εφαρμογή. Ανάλογα με τις τη κάθε κυβέρνηση. Πάση περιπτώσει όμως ε, μετά την μικρή ανάκαμψη του 2009 ε, στην οικονομική δραστηριότητα φαίνεται ότι αυτή η οικονομική κρίση απειλεί να μετατραπεί σε ένα τρίτο κύμα σε μια κρίση εξωτερικού χρέους, δημόσιου χρέους. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμη σε πλήρη ανάπτυξη, αλλά είναι πρώτον πυλών κατά την άποψή μου και το βλέπουμε ξεκάθαρα με την περίπτωση της Ιρλανδίας ότι δεν είναι καθόλου καθαρή εικόνα ως προς την χρέωση των κρατών των εθνικών προϋπολογισμών και γι' αυτό θα ήθελα να συζητήσω και το ζήτημα του ευρώ και της τάσης του κυρίου Φαν Ρόμποϊ. Εν πάση περιπτώσει όμως η δική μου έκθεση σχετίζεται μόνο με το 2009 όπου μπορούμε να πούμε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να εκτιμηθεί πως έχει αντιδράσει κατά τρόπο μετρημένο και μάλιστα ικανοποιητικό στην κρίση που είχε να αντιμετωπίσει. Διαφυλάσσοντας πολλές ε, οικονομικές δραστηριότητες και κλάδους από την κατάρρευση που όμως χρειάζεται να συνεχίσουν αυτές οι προσπάθειες έτσι ώστε να αναπτυχθούν στο μέγιστο δυνατό οι δυνατότητες ανάκαμψης με τα έκτακτα μέτρα κυρίως τα οποία έχει εισαγάγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το προσεκτικό ε, σχεδιασμό και την σταδιακή όταν έρθει η ώρα κατάρριξη αυτών των έκτακτων μέτρων ε, θα μπορέσει πιστεύω να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και αυτό που βλέπουμε ήδη τώρα στην Ιρλανδία και αλλού δείχνουν πόσο μεγάλη είναι η κίνδυνη. οποιαδήποτε παραβίαση των συνθήκων του ε, Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη που ήδη διαπιστώνεται θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπω αυτή που βλέπουμε ήδη στην περίπτωση τη Ιρλανδία και περαιτέρω πιθανέ παραβιάσει να αποτραπούν. Έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την εξισορρόπηση των οικονομικών στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών της ε, Ευρωζώνης και θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό διαχείρισης κρίσης στον οποίο θα μπορούμε να καταφύγουμε. Το ευρώ θα πρέπει να μετατραπεί σε έναν ασφαλή μηχανισμό για αποτροπή περαιτέρω κρίσεων. Η διαρθρωτική διαδικασία ανάκαμψη τη όνη του ευρώ νομίζω ότι δεν μπορεί παρά να ενισχυθεί με τα μέτρα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τη νέα διακυβέρνηση, οικονομική διακυβέρνηση και το νέο ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για, την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων. Ε, πιστεύω ότι έχουμε χρήσιμα εργαλεία στα χέρια μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο του τον εποπτικό και η κρίση πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά εφόσον όμως τους, προσεχείς, τους άμεσα προσεχείς μήνες μπορέσουμε να έχουμε μια σοβαρή στάση στην υπόθεση αυτή. Η κρίση αποτελεί όχι μόνο ένα κίνδυνο, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία ω εκ τούτου και γι' αυτό θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τι πολιτικέ ομάδε με τι οποίε συνεργάστηκα. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία. Δεν είναι ποτέ αυτονόητο κάτι τέτοιο και γι' αυτό το λόγο ήθελα ρητά να το αναφέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγική σα ομιλία. Θα ήθελα να καλωσορίσω στο Ευρωκοινοβούλιο τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο jean Jean-Claude Τρισέ. Κύριε Τρισέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, Herr Balt, αξιότιμο κύριε Ευρωβουλευτά, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με τη συνθήκη, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση για το 2009. Λόγω των ευρωεκλογών είχα μιλήσει εδώ το, πέρυσι το Μάρτιο. Είναι η δεύτερη φορά μάλλον φέτο το Μάρτιο ήταν οι ευρωεκλογέ, γι' αυτό είχε αλλάξει ημερομηνία και είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι ενώπιον σα και σα ευχαριστώ για την στήριξη μέσω του ψηφίσματο ε, υπέρ των, συνεχ... των τακτικών ακροάσεων ενώπιον της Επιτροπής ΕΚΟΝ και της στενής συνεργασίας με την ΕΚΤ. Χαίρομαι δε ακόμη παραπάνω για το γεγονός ότι φέτος το Ευρωκοινοβούλιο απέδειξε με πολύ δύναμη τη θέλησή του και την ικανότητά του να προασπίζεται το υπέρτατο συμφέρον της Ευρώπης όσον αφορά την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού πακέτου. Θα σας παρουσιάσω τώρα μια σύντομη επισκόπηση ως προς τις νομισματικές, τα νομισματικά μέτρα τα οποία εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Πέραν της χρονικής περίοδου της κρίσεως θα ήθελα να αξιολογήσω και την πρώτη δωδεκαετία λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και κλείνοντας θα ήθελα να ε, αναφερθώ στις ε, πλέον κατεπίγουσες ε, προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ή αναμένουμε να βρούμε μπροστά μας το 2011. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά την κρίση. Το 2009 ήταν ένα έτος πρόκληση για την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε με την παγκόσμια κρίση μετά από την το ξεκίνημα της χρημα οικονομικής ε, κρίσης το φθινόπωρο του 2008. Είχαμε πληθωριστικές πιέσεις, αλλά παρόλα αυτά συνεχίσαμε με την πολιτική μας να μειώνουμε ακόμη παραπάνω το επιτόκια μας. Και σε μία περίοδο μόνο 7 μηνών, μεταξύ Οκτωβρίου 2008 και Μαΐου 2009, <clears throat> μειώσαμε το επιτόκια μας κατά 325 πόντους και είμαστε τώρα στο 1%. Βεβαίως όλοι εποφελούνται στην στον ευρωπαϊκό χώρο από αυτές τις συνθήκες και, το 2009 συνεχίσαμε να υποστηρίζουμε τις ευρωπαϊκές τράπεζες με πιστώσεις. Αυτό λόγω της δυσλειτουργίας των αγορών, πράγμα το οποίο σήμαινε ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορούσε να επηρεάσει τη σταθερότητα με μόνο αποφάσεις για τα επιτόκια. Μεταξύ των μη σύνηθων μέτρων, το πιο σημαντικό είναι η ρευστότητα που δόθηκε μέσω της επαναχρηματοδότησης τραπεζών της περιοχής του ευρώ μέσω ασφαλιών για πολλές προθεσμίες οριμότητας που ξεπερνούν, ξεπερνούσαν ε, κατά πολύ την εβδομαδιαία ανανέωση. Επίσης το 2009 ανανεώσαμε αναχρηματοδοτήσεις για ένα έτος και αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Όπως σωστά το υπογραμμίζετε στο σχέδιο ψηφίσματος που έχετε, αυτή η υποστήριξη του δανεισμού βοήθησε να αποφύγουμε τυχόν πρόσθετες λειτουργίες που θα οδηγούσαν σε ύφεση πολύ χειρότερη. Θα ήθελα να σας πω ότι ευθυγραμμιζόταν όλες μας οι πράξεις με την μεσοπρόθεσμη προοπτική για τη σταθερότητα στην περιοχή του ευρώ. Μπορέσαμε αξιόπιστα να εκτελέσουμε την εντολή μας και βλέπετε ότι αυτό αντανακλάται από τον πληθωρισμό όπως εμφανίζεται ομαλά στην περιοχή του ευρώ. Μετά από κάποιες βελτιώσεις στις αγορές το 2009, στη συνέχεια αντιμετωπίσαμε νέες εντάσεις για τα ομόλογα στην περιοχή του ευρώ πάντοτε. Η ομαλή λειτουργία της αγοράς των ομολόγων είναι πολύ σημαντική για τα κεντρικά επιτόκια της ΕΚΤ. Γι' αυτό παρέμβημεν για να αποκαταστήσουμε μια πιο ομαλή ε, νομισματική πολιτική σε σχέση με την οικονομία. Εισαγάγαμε λοιπόν το σύστημα ασφάλιων, νομισματικών ασφαλιών και, γεννα... και ξανααπορροφούμε όλη την ρευστότητα που αρχικά δώσαμε για να μην επηρεαστεί η νομισματική μας πολιτική. Όλες οι ενέργειες οι μη που ε, πραγματοποιήθηκαν είναι προσωρινές στη φύση τους και σχεδιάστηκαν για να βγούμε από την κρίση. Ορισμένα μέτρα ξεκίνησαν την αρχή του 2009 και την αρχή του 2010 και ήδη έχουν ε, περατωθεί μετά τις βελτιώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την ανάκαμψη της σχετική της περιοχής του ευρώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω μερικές μου σκέψεις σε σχέση με την εξέλιξη του ευρώ. Τρία στοιχεία είναι θεμελιώδη. Πρώτα απ' όλα η ΕΚΤ έδωσε αυτό που έπρεπε να δώσει σύμφωνα με την εντολή που έχει από τις συνθήκες, δηλαδή σταθερότητα τιμών. Η μέση, ο μέσος πληθωρισμός στο ευρώ εδώ και 12 χρόνια είναι 1,97% πράγμα το οποίο αντανακλά τη σταθερότητα των τιμών και διατηρούμε ε, μέσο πληθωρισμό στην περιοχή του ευρώ κάτω από το 2 και πολύ κοντά στο 2. Με από αυτή την άποψη το σύστημα του ευρώ τα τελευταία 12 χρόνια έχει λειτουργήσει σαν άγκυρα σταθερότητας και εμπιστοσύνης ακόμη και στους πολύ πρόσπατους καιρούς παρά τα γεγονότα τα οποία προκλήθηκαν από την παγκόσμια κρίση. Δεύτερον, επηρεάζει θετικά την νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, δηλαδή οι πληθωριστικές τάσεις έχουν ευθυγραμμιστεί με τη σταθερότητα των τιμών. Τρίτον, η επιτυχία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανεξαρτησία της ΕΚΤ από τις πολιτικές δυνάμεις για και γι' αυτό μπορεί και διατηρεί σταθερότητα τιμών και έχει διαφανή επικοινωνία σε αυτούς τους τομείς. Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ μας επιτρέπει να είμαστε ε, προσανατολισμένοι μεσοπρόθεσμα με βάση ένα σταθερό πλαίσιο αναλυτικό το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις τις νομισματικές και τις πιστοτικές ε, από το μεσοπρόθεσμο μέχρι το μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να είμαστε ενημερωμένοι στις αποφάσεις μας και συνεπείς στη γραμμή μας, σταθεροί, ώστε να αποφεύγουμε την πτυτικότητα, αν θέλετε, την στιγμιαία. Επίσης, το νόμισμά μας έχει εγκαθιδρυθεί παγκοσμίως το 2009 αντιπροσώπευε το 30% των ασφαλιών για πιστώσεις και των αποθεμάτων. Όσον αφορά τώρα την εξωτερική πτυχή του ευρώ, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα συναλλαγματικά. Ε, θα έλω να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε αυτούς τους τομείς. Υπάρχουν δύο βασικά θέμα, θέματα, η σχέση μεταξύ των μετατρεψίμων ε, νομισμάτων των βιομηχανικών χωρών ε, ε, ευρώ, καναδικό δολάριο, δολάριο ΙΠΑ, λίρα, μετά την κατάρρευση του συστήματος του Bretton Woods, αυτά τα νομίσματα κυμαίνονται. Και η υπερβολική πτυτικότητα και η αταξία, αν θέλετε, στις κινήσεις τις συναλλαγματικές έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην οικονομική σταθερότητα και την νομισματική. Η ΕΚΤ πρέπει να σας πω ότι χάρη και για τις πρόσφατες δηλώσεις των Αμερικανικών αρχών του Υπουργού Οικονομίας και του Προέδρου του Federal Reserve. Δηλαδή είπαν ότι η σταθερότητα είναι προς όφερος, τον είπα και βεβαίως συμφωνώ ότι ένα δολάριο το οποίο είναι αξιόπιστο είναι προς συμφέρον τον ΗΠΑ, της Ευρώπης και όλης της παγκόσμιας κοινότητας. Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω είναι οι αναδυόμενες οικονομίες και τα νομίσματά τους. Έχουν συναλλαγματικές ισοτιμίες που δεν είναι επαρκώς ευέλικτες. Πάνω σε αυτό το θέμα η διεθνής κοινότητα συμφωνεί και ελέγχθη αυτό και την περασμένη εβδομάδα άλλωστε ότι η κίνηση προς μια συναλλαγματική πραγματικά αγορά και η αποφυγή υποτιμήσεων για λόγους ανταγωνιστικούς είναι προς συμφέρον των αναδειωμένων οικονομιών και της παγκόσμιας κοινότητας. Λοιπόν κύριε Πρόεδρε, η ΕΚΤ έλεγε ότι δεν είναι καιρός τώρα για να εφησυχάζει κανείς. Πράγματι, έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας Όλες οι αρμόδιες αρχές γνωρίζουν τα θέματα του ιδιωτικού τομέα, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, έχουμε τις ρυθμιστικές αρχές, τον ιδιωτικό τομέα και την χρηματοοικονομική αγορά. Λοιπόν, η κρίση η τρέχουσα έχει αποδείξει ότι η εφαρμογή θαραλέων μεταρρυθμίσεων είναι προς συμφέρον και των χωρών του ευρώ και του ευρώ στο σύνολό του. Η πρόταση του Προέδρου Φων Ρόμπο για τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης και τη η έγκριση από το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2010 αντανακλούν μια βελτίωση στο ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι σκόπιμο, είναι χρήσιμη και για τις χώρες ε, της Ευρώπης, τα χώρες μέλη που δεν συμμετέχουν στο ευρώ αλλά από την άλλη πλευρά είναι λιγότερες από αυτό που απαιτείται για να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη λειτουργία του ενιαίας, ε, της οικονομίας με ένα ενιαίο νόμισμα. Είμαι σίγουρος ότι τους επόμενους μήνες το Ευρωκοινοβούλιο θα βοηθήσει την Ευρώπη να κάνει το σημαντικό βήμα προς την ε, οικονομική διακυβέρνηση. Έχετε υποπτικό ρόλο και πρέπει να καταδείξετε την αποφασιστικότητά σας όταν πρόκειται για κέρια θέματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την τοποθέτησή σας και θέλω και πάλι να σας πω ότι θα είναι σημαντική η επίδραση του Κοινοβουλίου στη συζήτηση για τη διακυβέρνηση. Ένα άλλο σημαντικό θέμα έχει να κάνει με τις χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις. Πρέπει να διατηρήσουμε την ε, ενέργεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή για μια τέτοια μεταρρύθμιση και μάλιστα γρήγορα. Η νομοθετική πρόταση για το short selling και για άλλες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες να προχωρήσουν για να γίνει πιο διαφανές το σύστημα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τι αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης. Αντιμετωπίζουμε μια σημαντική χρονιά. Το 2011 πρέπει να οδηγήσει στη μεταρρύθμιση σε βάθος του πλαισίου λειτουργίας και να ξεκινήσει ενδεχομένως και η διαδικασία για τη τροποποίηση της συνθήκης. Οι μεταρρυθμίσεις όλες πρέπει να γίνουν σωστά ώστε η Ευρώπη στο σύνολό της και η περιοχή του ευρώ ειδικότερα να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη αξιοπιστία και πεποίθηση στο μέλλον. Και όπως λέτε στο σχέδιο ψηφίσματός σας, κάνουμε το βέλτιστο που μπορούμε για να υποστηρίξουμε την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια της ΕΚΤ. Έχω ήδη ε, μιλήσει για αυτό το σημαντικότερο θέμα κατά το παρελθόν στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα συνεχίσουμε να εκτελούμε την εντολή μας, αυτό ζητάει συνθήκη από εμά και πιστέψτε με θα προχωρήσουμε όπως το αναμένουν οι πολίτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ομιλία σας. On behalf of the European... Εκ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος, ο κύριος Ρεν. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αξιότιμα μέλη, καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Μπούρχαρτ Πάλτς, για την πολύ αναλυτική του την πληρέστατη έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται αυτή την έκθεση που αντικατοπτρίζει με σωστό τρόπο τα βασικά θέματα που τίθενται η έκθεση αναγνωρίζει και εκτιμά το έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην διαχείριση της κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με αυτή την άποψη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπό την ηγεσία του Προέδρου Jean-Claude Trichet πλοήγησε εν μέσω της δυσκόλου αυτής καταστάσεως με θεπιδεξιότητας, με σταθερό χέρι. Και δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω τον Jean-Claude Τρισέ για την έξοχη συνεργασία και σας ευχαριστώ κυρίως για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίσατε αυτή την περίοδο των αναταράξεων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της νομισματικής τοποθέτησης και των ειδικών μέτρων διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να ξεπεραστεί η κρίση, στην πυρόσβεση της κρίσης και έθεσε τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η έκθεσή σας σωστά υπογραμμίζει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη για ενισχυμένη οικονομική εποπτεία και έλεγχο στην Ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με αυτό. Ακριβώς γι' αυτό υποβάλαμε διάφορες προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβερνήσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερο στην Ευρωζώνη. Επίσης λάβαμε υπόψη μας αρκετές προτάσεις που υποβλήθησαν στην έκθεση ΦΕΙΟ για την ενίσχυση της ε, οικονομικής διακυβερνήσεως στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Οικονομική Επιτροπή ε, παρέλαβε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κινείται Προ την φιλόδοξη προθεσμία του Ιουνίου του επομένου έτους να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αυτό είναι ευπρόσδεκτο, αυτός ο στόχο. Στρέφομαι τώρα στο δεύτερο τμήμα της συζητήσεώ μας που αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τις διεθνείς ισοτιμίες. Σωστά αναφέρεται ότι η πτητικότητα των αγορών ξένων συναλλαγμάτων αυξήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες με σημαντικές μεταβολές όσον αφορά τις ισοτιμίες των διαφόρων, τις διάφορες ισοτιμίες μεταβλήθηκαν σημαντικά. Το ευρώ ανατιμήθηκε έναντι του δολαρίου από τον Ιούνιο και πέρα λόγω ε, καλυτέρων στοιχείων για την οικονομία της Ευρωζώνης και λόγω ε, και ε, της νομισματικής πολιτικής που ακολούθησαν οι ΕΠΑ. Όμως, πρόσφατα, το ευρώ αδυνάτησε έναντι των περισσότερων ε, νομισμάτων και αυτό αύξησε τις ανησυχίες για τα δημοσιονομικά των κρατών μελών και πάνω απ' όλα στην Ιρλανδία. Και οι ανησυχίε, για, για διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων και η Ιρλανδία επηρέασε το ευρώ. Στην πραγματικότητα το ευρώ είναι στο, κοντά στο μακροπρόθεσμο μέσο όρο τη τιμή του λαμβάνοντα υπόψη και τι διάφορε υποτιμήσει που έγιναν φέτο, ενώ πέρσι ήταν υπερτιμημένο. Οπότε ο μέσο όρο είναι κανονικό. Εν συγκρίση με τι αρχέ του έτου, η υποτίμηση του ευρώ σε πραγματικού όρου είναι περίπου 7%. Στα πλαίσια της αργής ανακάμψεως στις προθυμένες οικονομίες και τις μεγάλες κεφαλαιακές ροές στις αναδιόμενες οικονομίες, Πολλές χώρες προσπαθούν να υποτιμήσουν το νόμισμά τους ή τελικά καταπολεμούν ε, την αύξηση της αξίας του νομίσματός τους. Και θα πρέπει, και γι' αυτό οι ηγέτες των G20 Σεούλ την περασμένη εβδομάδα πολύ ξεκάθαρα δεσμεύτηκαν να πόσχουν από ανταγωνιστική υποτίμηση των νομισμάτων τους. Η G20, η Σύνοδος Κορυφής των G20, οδήγησε μια συμφωνία. Προσπάθησαν να, εξι... να γίνουν προσπάθειες για επανεξισορρόπηση της παγκόσμιας ανάπτυξης. Κατέληξαν σε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Ευελιξία όσον αφορά τις ισοτιμίες πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο για την επανεξισορρόπηση των οικονομιών, ούτω ώστε η ισοτιμία να αντικατοπτρίζει τι βασικέ οικονομικέ αρχέ. Κάτι που ανέφερε και ο πρόεδρο ο κύριο Τρισέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει την υποστήριξη τη σημαντική προσπάθεια που κάνουν οι G20 και εκεί θα εστιαστεί και η Γαλλική Προεδρία των G20 το επόμενο έτος. Τέλος, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, πρέπει να σας ενημερώσω για κάτι Έχαμε σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την Ευρωζώνη χθες στο Συμβούλιο Κοφίν έγινε δεκτή η αίτηση της Ιρλανδικής κυβερνήσεως για οικονομική ενίσχυση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Υπουργοί συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι η παροχή βοηθείας στην Ιρλανδία απαιτείται για να διαφυλαχθεί η οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη. Η οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορεί να παρασχεθεί μέσω ενός προγράμματος με αυστηρούς όρους πολιτικής, κάτι που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης τώρα με τις ε, αρχές της Ιρλανδίας. Γίνονται διαπραγματεύσεις με συμμετοχή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα, θα προσπαθεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της Ιρλανδίας με αποφασιστικό τρόπο και το πρόγραμμα αυτό θα συμπεριλαμβάνει και ένα ταμείο για ενδεχόμενες μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα και για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των τραπεζών προβλέπονται διάφορα μέτρα όπως αναδιάθρωση και μόχλευση της οικονομίας ούτως ώστε τελικά το τραπεζικό σύστημα της Ιρλανδίας να παίξει το ρόλο του όπως πρέπει στα πλαίσια της γενικότερης οικονομίας. Οι συνομιλίε τεχνικού περιεχομένου που αφορούν το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Νομισματικού Ταμείου έχουν ξεκινήσει και οι διαπραγματεύσει ίσω να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλο του Νοεμβρίου. Πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Διεθνού Ταμείου και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία ανέφεραν, δήλωσαν ότι είναι έτοιμες αυτές οι δύο χώρες να συμβάλλουν στο πρόγραμμα μέσω διμερών δανείων και αυτό είναι πρόσδεκτο. Εν γέννη, οι χθεσινέ αποφάσεις είναι ένα κρίσιμο βήμα προόδου όσον αφορά τις κοινέ προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της Ιρλανδική οικονομίας και έτσι να διαφυλαχθεί η οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος, για την εισαγωγή που κάνατε στο θέμα αυτό. Ε, εκ μέρους των πολιτικών ομάδων τώρα. Εκ μέρους του ΕΛΚ, ο Ζαν Πολ Γκοζές έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα συμφωνήσω και εγώ βεβαίως με όλους τους επένους που ακούστηκαν για τι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν θα επαναλάβω τα λόγια του κυρίου Μπάλτ για τα όσα έχουν περιληφθεί μέσα στο ψήφισμα. Έχω πολύ λίγο χρόνο στη θέση μου και γι' αυτό θα ήθελα απλώ να σα πω ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε τον συμπολίτη μα, να σκεφτούμε τον συμπολίτη μα. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί χθε το βράδυ κάθε ε, ραδιοτηλεοπτικό σταθμό στη Γαλλία είχε και από έναν υποψήφιο ε, στις μελλοντικέ προεδρικές εκλογές, ο οποίος ε, κατέβαινε για να, δείξει, να δείξει ότι καταστρέφει από τη ρίζα το κακό ε, και έτσι έσκιζε μπροστά στην κάμερα ένα φωτοαντίγραφο ε, νομίσματος, χαρτονομίσματος των 10 ευρώ. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι δεν είναι εκεί το ζήτημα, ούτε έτσι λυνώζονται τα προβλήματα. Η εποπτεία, η ο αυστηρός έλεγχος που αναφέρατε και εσείς κύριε Πρόεδρε είναι ακριβώς ε, απαραίτητη αλλά ταυτόχρονα πρέπει και αυτή είναι η δουλειά του Κοινοβουλίου να εξηγήσουμε στο συμπολίτη μας μηνύματα τα οποία δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί γιατί διαρκώς παρουσιάζονται από τον τύπο διάφορες ε, εικόνες ε, δυσνόητες για τον πολίτη ε, καταστάσεις πολύ δύσκολες και προχτές που συναντήθηκα με συμπολίτε μου, άκουσα από το στόμα του ερωτήσεις σχετικέ με την Ευρωζώνη και το ευρώ. Φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνονται πόσο καλή είναι η δουλειά τη Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ από τους σοσιαλιστέ και δημοκρατικούς, ο κύριος Τζορτ Σαμπιν Τσούτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Τρισέ, κύριε Ρέν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάλτς για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και να χαιρετήσω το ιδιαίτερο καθεστώς ε, που αποδόθηκε από τη συνθήκη της Λισαβόνας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα ήθελα επίσης ε, να ε, καταγγείλω σημαντικές αποκλήσεις στα επίπεδα τα οικονομικά μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται πιο στενές ε, οικονομικές και νομισματικές πολιτικές. Δεν αρκεί ανάπτυξη μόνο για να καλυφθούν τα μεγάλα χάσματα, οι μεγάλες αποκλήσεις οικονομικές μεταξύ των κρατών. Πρέπει να δοθεί με έναν μηχανισμό αλληλεγγύης η ευκαιρία της έκδοσης Ευρώ ομολόγων, Έτσι, εκείνη η χώρα η οποία θα βρίσκεται σε δυσκολία θα μπορεί να ε, βοηθηθεί ενισχύοντας ταυτόχρονα και τη δυνατότητα ε, δημοσιονομικής εποπτείας αλλά και εξασφαλίζοντας προς τη ρευστότητα. Πρέπει λοιπόν μαζί με το ευρώ να εξασφαλιστεί και η δημοσιονομική αυστηρότητα, η τήρηση δηλαδή, των ε, δημοσιονομικών διατάξεων και η εποπτεία. Η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση έχει συγκλονίσει, έχει ε, κλειδονίσει πολλές οικονομίες ευρωπαϊκές και επιπλέον κερδοσκοπικές επιθέσεις κατέστησαν πολύ πιο δύσκολο το δανεισμό των κρατών αυτών στις διεθνείς αγορές. Εδώ χρειάστηκε να αναλάβει δράση λοιπόν η Ευρωζώνη και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα μόνιμο μηχανισμό που θα προστατεύει το ευρώ από τις κερδοσκοπικές επιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Τρικεντρική Τράπεζα πιστεύουμε θα πρέπει να αναλάβει την εποπτεία, τη διαχείριση των ε, οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ε, ικανότητας και ίσως να είναι σκόπιμο να θεσπιστεί και ένας ευρωπαϊκός τέτοιο οργανισμός. Έτσι θα μπορέσουμε πιστεύω να δούμε την ανάκαμψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ένα ευρωπαϊκό σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης με δημοσιονομική ενοποίηση που θα οδηγεί σε με μάλλον ενίσχυση των οικονομικών να οδηγήσει και σε νέες θέσεις εργασίας και με κάλυψη των μεγάλων χασμάτων μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών και φυσικά με πράσινη οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκουλάρ, από τους φιλελεύθερους και δημοκρατικούς του Κοινοβουλίου. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε της Τράπεζας. Καταρχάς, και εγώ θέλω να επενέσω τον εισηγητή μα, ο οποίος νομίζω ότι καλά στόχευσε όσον αφορά το θέμα. Στην έκθεσή του υπογραμμάζει τις καινοτομίες που επέφερε η συνθήκη Λισαβόνα και θα ήθελα πραγματικά να σε ευχαριστήσω κύριε Τρισέ που το υπενθυμίσατε αυτό απόψε. Ε, σε εκείνου που τα γνωρούσαν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που υπέγραψαν και επικύρωσαν τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η συνθήκη αυτή τη Λισαβόνα φέρνει μια μεγάλη καινοτομία. Θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε δημοσία σε αυτό το χώρο όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση του φόρου Σταθερότητα υπό την ευθύνη του κυρίου Ρεν, έδωσε μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διάφορα κείμενα που ακολουθούν την σωστή κατεύθυνση, αρκετά θαραλέα και θέλουν να δυναμώσουν την πειθαρχία, ζητώντα να ληφθούν υπόψη οι ανισορροπίε οι μακροοικονομικέ που ο κύριο Μπάλτ ανέφερε και εκείνο στην έκθεσή του. Και αναφέρεται κύριο Τρισέ επανειλημμένα στα γαλλικά ένα κβαντικό άλμα ε, όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Ε, ομολογώ ενώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο Ζαν Πολ Γκαζές, ότι όταν πηγαίνουμε επί τόπου, διερωτώμεθα κατά πόσο αυτές οι προτάσεις οι οποίες έγιναν το Σεπτέμβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επίκαιρε. Μήπως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κρίση η οποία σοβεί σε αυτή τη φάση, ούτω ώστε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Και θέλω να επιθυμίσω εδώ ότι που, εκείνοι που συνέλαβαν τη ιδέα του ευρώ δεν φανταστήκαν ποτέ ότι θα είχαν μια απλή, ε, ένα απλό συντονισμό οικονομικών πολιτικών μακροπρόθεσμα. Είχαν υπόψη τους μια οικονομική ένωση, δηλαδή μια δυνατότητα ε, λήψης αποφάσεων ε, υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Αυτό που με εκπλήσει κάπως για να αναφερθώ και στους πολίτες, είναι ότι έχουμε αυτοκινητιστές, τα κάτι μέλη, που καμιά φορά είναι στο τιμόνι ε, και μετά ε, και τους ίδιους βάζουμε και στην άκρη του, του διαδρόμου να κάνουμε να κόβουν τα πρόστιμα. Ε, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει μια χώρα στην οποία η κυκλοφορία στο δρόμο γίνεται με αυτόν τον τρόπο δηλαδή και ελέγχοντε και ελεγχόμενοι να είναι οι ίδιοι, θα πρέπει να αυξήσουμε και τα πρόστιμα και καλά κάνατε που υπενθυμίσατε ότι κάναμε κάτι για την προάσπιση των, ε, του χρηματοστατικού τομέα και για τον, χρηματοστατικό, τον έλεγχο του χρηματοστατικού τομέα. Ευχαριστώ πολύ κυρία. Λοιπόν, ο κ. Σβέν Γκίγκολτ ε, για τους πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, από πλευρά μας και για τον ε, κύριο Μπάλτς για την εξαιρετική συνεργασία. Ήταν μια πολύ καλή έκθεση, ισορροπημένη. Το 9 και το 10 ως έτη χαρακτηρίζονται από τα έκτακτα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εν ώψη των όλων εξαιρετικών οικονομικών εξελίξεων έλαβε αυτά τα έκτακτα μέτρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και θα ήθελα ρητά να ευχαριστώ τον κύριο Τρισέ για την προσπάθειά του, η οποία ξέρω ότι ήταν και αρκετά ε, ακανθώδης. Δεν ε, βρήκε πάντα ευήκοα ότα όταν θέλησε να επιβάλλει τα μέτρα αυτά. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πολιτική η οποία θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το, εξωτερικό, το δημόσιο χρέος αλλά και το ιδιωτικό, μια πολιτική η οποία θα στρέφεται και προς τα κράτη τα ελληματικά αλλά και προς τα κράτη που παρουσιάζουν πλεονάσματα και που θα εξετάζει και τις τιμές καταναλωτού αλλά και την αξία των περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να οδηγούν σε ε, κερδοσκοπικές πιέσεις και φούσκες. Ταυτόχρονα όμω χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο για τον φορολογικό ανταγωνισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν προγράμματα λιτότητας σε ορισμένα κράτη, τα οποία όμως ταυτόχρονα χάνουν ε, τα φορολογικά έσοδα που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν λόγω του φορολογικού ανταγωνισμού, θέμη του ανταγωνισμού από κάποια άλλα. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε σήμερα να διασώσουμε τις τράπεζες της Ιρλανδίας, μεν χωρίς όμως να πιέζουμε για την αύξηση του ε, κατά τρόπο σκανδαλώδη χαμηλό, χαμηλού ε, φόρου για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που είναι στο 12% και δεν λέμε τίποτα για το γεγονός ότι θα έπρεπε αυτός να ανέλθει στο 25% όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ταυτόχρονα, λοιπόν, θα ήθελα να επισημάνω ότι ήταν ε, καλό να μας πείτε μερικά πράγματα πιο συγκεκριμένα για τις ε, ασφάλειες, για τις εγγύησεις. Ε, πιστεύω ότι μιλάω εκ μέρους όλων των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ η κυρία Σουίνμπερν από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μπάλτση την έκθεσή του. Τη στιγμή όμως ε, που αντιμετωπίζει καθημερινές πιέσεις και κρίσεις το ευρώ και που αναφέρει το χρειάζονται νέοι κανόνε και νέα διακυβέρνηση για την ε, επιβίωση του, πώ είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στέκεται έξω από τι παγκόσμιε εξελίξει. Εδώ έχουμε του ε, μεγάλου παγκόσμιου ε, παράγοντε που υποχρεωμένοι πλέον να συνεργαστούν, να αναζητούν λύσει για την αντιμετώπιση τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Μια μεταρρύθμιση ως προς την οικονομική διακυβέρνηση και κυρίως ε, των χρηματοπιστωτικών παραγόγων κατέστη απαραίτητη ή μεγάλη κλειδονισμή που υφίστανται οι διεθνείς, ε, οι παγκόσμιες, οι διεθνείς τράπεζες, οι πολυεθνικές τράπεζες θα μας υποχρεώσουν να λάβουμε δράση. Υπάρχει από τη μια πλευρά όμως η Fed η οποία προσπαθεί να διαφυλάξει, να προστατεύσει το δολάριο, από την άλλη οι Κινέζοι προσπαθούν να προστατεύσουν το Ιουάν και ίσως εμείς να βρεθούμε επί ξηρού κρεμάμενοι στην υπόθεση αυτή. Και πιστεύω ότι παρά τι εσωτερικέ, έντονε εσωτερικέ πιέσει, μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί έχει και τη σχετική ε, γνώση και ε, ε, πραγματογνωμοσύνη στην υπόθεση αυτή, να πιέσει στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κλούτε, εκ μέρου τη Νομόσπονδη τη Ομάδα τη Ευρωπαϊκή Αριστερά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον συνάδελφο Μπάλτσα για την πολύ καλή συνεργασία. Δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω ότι και τη δική μα έποψη ήταν πολύ καλή συνεργασία. Πολύ θεωρούσαν ότι η κρίση της ζώνης του ευρώ είχε πια παρέλθει, όμως η Ιρλανδία αποδεικνύει με την περίπτωσή της ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υφίστανται σημαντικές πιέσεις από τις χρονοπετσοστικές αγορές εις βάρος των ευρωπαϊκών κρατών. Αναγκάζεται η Ιρλανδία να εκτεθεί στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές ε, ζητώντας ε, ελεημοσύνη με πολύ ψηλά επιτόκια, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλει ε, πολύ σκληρά μέτρα λιτότητας. Αυτό που είδαμε δηλαδή και με την Ελλάδα βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και στην Ιρλανδία με ταυτόχρονα όμως προσπάθεια προστασίας και διάσωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ενώ πρώτον πυλών έρχεται η ε, συνθηκολόγηση της πορτοκαλίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν σε αυτής της δραματικής και τραγικής καταστάσεως έχει προτείνει μια εναλλακτική ε, η οποία ισοδυναμεί λίγο πολύ με ένα κρατικό καζίνο οδηγεί δηλαδή την κάθε χώρα με τις πιεστικές της και πολύ αυστηρές ε, τα πολύ αυστηρά της μέτρα και την πιεστική της πολιτική στην φτώχεια, στην εξαθλίωση και θα έλεγα κύριε Τρισό ότι είναι καλό να κοιτάξετε την αλφαβήτα της οικονομίας για να καταλάβετε ότι τα κρατικά ομόλογα δεν μπορούν να μένουν στον αέρα, πρέπει να προστατευτούν και πρέπει να προστατευτούν οι εθνικές οικονομίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλούτε. Υπάρχει μια συμπληρωματική ερώτηση για τις δηλώσεις από τον κύριο Χάνς Πέτερ Μάρτιν. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε να γίνει συζήτηση. η ανταλλαγή μάλλον. Δεν έχω αντίρρηση, λέει ο κύριο Κλούτε. 30 δευτερόλεπτα, κύριε Χάνι Πέτερ Μάρτιν, για να δοθεί μετά η απάντηση. Κύριο Χάνι Πέτερ Μάρτιν, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κλούτε, τον συνάδελφο. Αυτό που προτείνει, η συνταγή που έχει υπόψη για οργανωμένα ευρωομόλογα, ευρωπαϊκό δανεισμό. Σε ποιο βαθμό είναι συμβατά με τις σχετικές αποφάσεις του, του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ομοσπονδιακού Σταγματικού Δικαστηρίου. Και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα προκύψουν στη συνέχεια αποφάσει του Ευρωπαϊκού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, Συνταγματικού Δικαστηρίου τη Καρλσρούη, ε, που θα ανατρέψουν τέτοιε περιπτώσει, κύριο Κλούτε. Ε, ομολογώ ότι είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανεί αυτήν την κατάσταση. Είναι δύσκολο βεβαίω. Από την άλλη όμω έχει προχωρήσει τόσο πολύ η κατάσταση που ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε και τρόπο θεώρησης όλης αυτής της οργάνωσης. Αλλά εύκολη απάντηση στην ερώτηση σας δεν έχω δυστυχώς. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Συνεχίζουμε με τους ε, ομιλητέ με τη σειρά όπως τους έχουμε. Ο κύριος Μπάφτον καταρχάς, Ευρώπη των Ελευθεριών και των Δημοκρατιών. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε διάβασα την έκθεση της Επιτροπής της Νομισματικής και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την έκθεση της και είναι πολύ ενδιαφέρον, λέει ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών της Ευρωζώνης και αυτό συνέβαλε στα προβλήματα που βλέπουμε σήμερα. Η έκθεση αναφέρει ότι είναι ανισορροπίες που δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τη σωστή νομισματική πολιτική εντός της Ευρωζώνης και επαναλαμβάνει ότι η χρηματοστατική κρίση σε κάποιες χώρες είναι ένα σοβαρό θέμα για τον γενικότερο τομέα και αντικατοπτρίζεται μέσω της λειτουργίας Ευρωζώνης. Εγώ δεν βλέπω τι νομο υπάρχει να μιλάμε για μεγαλύτερο συντονισμό οικονομικών πολιτικών εντός Ευρωζώνης. Η άμεση αντίδραση ήταν η αύξηση της οικονομικής διακυβέρνηση, αλλά είναι περιορισμής οι περιορισμοί και επιβεβλημένη κοινή προσέγγιση που οδήγησε στην οικονομική κρίση με εξωτερικούς λόγους που είναι ανεξέλεγκτοι. Ίσως ένα σύστημα δεν επιτρέπει την αναγκαία οικονομική ελαστικότητα και αυτοκαθορισμό, τόσο ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα διάφορα ε, προβλήματα, τα ιδιαίτερα όπως είναι ο πληθωρισμός. Το τονίζει αυτό η έκθεση και σημειώνει ότι η κρίση και μετά οι προσπάθειε διασώσεω και των όσων οικονομία οδήγησαν σε πολύ αυστηρά μέτρα λιτότητα που περιορίζουν πάρα πολύ τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να κινηθούν και να δράσουν. Ένα επιχείρημα είναι ότι δεν μπορεί κανεί να έχει ένα νέο νόμισμα χωρί να εξομαλεί διαφορέ μεταξύ κρατών μελών και επίπεδου πλούτου. Όμω οποιοδήποτε ρεαλιστή γνωρίζει ότι κάτι δεν μπορεί να συμβεί. Είναι αντίθετο με την ανθρώπινη φύση. Που λογικά θα πρέπει αυτό να προβάλλεται σε μια οικονομία όσο και αν δημιουργεί προβλήματα. Είναι έτοιμη για την Εστονία τον Ιανουάριο Ευρωζώνη. Εγώ σηκώνω τα φρύδια μου βλέποντα τη δήλωση εθέτηση του νομίσματο από την Εστονία. Δείχνει ότι το καθεστώ του ευρώ είναι καλό και θα πρέπει και άλλα κατημέλη να μπουν. Η ιδεολογική προσκόλληση στην Ευρωζώνη ε, είναι κάτι που μας δημιουργεί προβλήματα. Το νέο νόμισμα ε, λειτουργεί μόνο σε ομοσπονδιακό περιβάλλον, πολύ αυστηρό. Ίσως αυτή να είναι τελική πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό τελικά κάνουν, ε, δημιουργούν προθύστερα. Παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι στην Ευρωζώνη, εμείς υποφέρουμε λόγω των προσπαθειών διάσωσης και λόγω της αλληλένδετης οικονομίας της Ένωσης. Άρα δεν έχει νόημα να περιμένουμε τη στιγμή που θα πούμε να είχαμε δίκιο. Πέρασε αυτή τη στιγμή που μπορούσαμε να πούμε ότι είχαμε δίκιο. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων, ο κύριος Χάνης Πέτερ Μάρτιν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μακάρι να μπορούσαμε να εγκρίνουμε την έκθεση του κυρίου Μπάλτσα ή να την σημειώσουμε με ένα υπόμνημα, θα έλεγα με ένα προσυπόμνηση. Κύριε Τρισέ, εσείς όσοι θα μπορούσατε να κάνετε μια αναδρομή στις εκθέσεις του 2008-2009, γιατί ορισμένους έχουμε να κάνουμε με ένα ταξίδι πάνω στα σύννεφα, πάνω σε ένα ρόδινο συννεφάκι. Υπάρχει λοιπόν η πρόταση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και του κυρίου Τρισέ για παράταση των αυτών μέτρων που φαίνεται ότι είναι καλά. Θα δούμε. Α μην ε, ε, κατηγορούμε αυτομάτως όλοι τον Greenspan. Αλλά το βασικό και το πιο αμφίβολο από όλα είναι ότι ο πολίτης δεν γνωρίζει όλα αυτά τα χρήματα, όλη αυτή η ρευστότητα που πάει και ότι όλη αυτή η ασπίδα προστασίας ή η ομπρέλα προστασίας η οικονομική διατίθεται κατά τρόπο τελείως αδιαφανή. 35 δισεκατομμύρια από τα ε, κονδύλια τα οποία πηγαίνουν στην Ιρλανδία ε, πάνε σε μια θηγατρική της γερμανικής Hippo Real Estate. Ποιος είναι εδώ πέρα ο μηχανισμός και ποιον διασώζουμε τελικά. Μια γερμανική τράπεζα, μια Ιρλανδική τράπεζα, το Ιρλανδικό κράτος πρέπει να είμαστε θέση να πούμε στον πολίτη αυτός τον οποίο θέλουμε να σώσουμε είναι ο τάδε, ο δίνα, αυτά τα χρήματα του δίνουμε και έτσι μόνο μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα της κατάστασης μέσα στην Ιρλανδία. Και επίσης το Ιρλανδικό τραπεζικό σύστημα που σε τελευταία ανάλυση είναι και υπέτειο για αυτή την κρίση. Γιατί να μην είμαστε αρκετά θαραλέοι ώστε να δεχθούμε και το ενδεχόμενο μια χρεοκοπία, μια πτώχευση μια Ιρλανδική τράπεζα, όπω συνέβη και με του Lehman Brothers, για να αλλάξουμε τα μερικά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Θα δούμε μετά του ομιλητέ, ε, ξεδιονόματο. Γκάλ Πέλτ, καταρχά. Θα ήθελα καταρχάς, Πρόεδρε, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον εισηγητή, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μην ξεχνάμε ότι είναι το ε, όργανο εκείνο το οποίο μπορεί να καλέσει λογοδοσία την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενώπιον των πολιτών της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τρισέ και που ήρθε εδώ σήμερα, αλλά περισσότερο που έχετε τακτικά και αναπτύσσει μεταξύ, ε, μεταξύ ημών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυτόν τον διάλογο για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τη ζώνη του ευρώ. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη και παγκόσμια ευθύνη δεν πρέπει να λησμονούμε το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη έχουν και χρηματοπιστωτικά και οικονομικά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Συμφωνώ με τον συγητή ότι τα κράτη-μέλη δεν εκλήθησαν να τηρήσουν με αυστηρούς όρους το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και εκεί εντοπίζεται η ρίζα του κακού. Μπορούμε να οδηγηθούμε δε σε ένα τρίτο κύμα κρίσεως που θα είναι η κρίση δημοσίου χρέους. χρέους. Ε, βλέπω με ικανοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιδρά με θετικό τρόπο, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται μια οικονομική ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ενισχύει και την, Ευρω... και την νομισματική ένωση, την Ευρωζώνη δηλαδή. Πιστεύω ότι θα πρέπει πάνω απ' όλα να διδαχθούμε από την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέμπελς για τρία λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετατρέψιμα νομίσματα δεν έχουμε μετά από την τρελή οικονομική κρίση. Το χρέος των κρατών είναι σοβαρό το πρόβλημα. Όμως η κρίση οφείλεται στη διάσωση ιδιωτικών τραπεζών. Η χρηματοπιστωτική κρίση επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στην πραγματική οικονομία. Μείωσε τις ε, δραστηριότητες και αύξησε την ανεργία οι επιζήσαντες του Wall Street, της Wall Street και της City <clears throat> κερδοσκοπούν και πουλάνε ε, υποτιμημένα τα CDS τα οποία δεν έχουν καν στα χέρια τους. Και κινδυνεύουν κράτη διότι εφαρμόζουν λιτότητα που θα καθιστά την ανάκαμψη πολύ, ε, πολύ πιο δύσκολη. Η αλληλεγγύη ευρωπαϊκή είναι ελάχιστη. Η διάσωση της Ελλάδας πρώτο απ' όλα σημαίνει διάσωση γαλλικών και γερμανικών τραπεζών. Η υποστήριξη της Ιρλανδίας σημαίνει διάσωση βρετανικών τραπεζών <clears throat> που θα υποφέρανε πάρα πολύ από την κατάρρευση των Ιρλανδικών τραπεζών. Το γεγονός ότι η ε, ισοτιμία του ευρώ κυμαίνεται, αυτό δεν είναι αδυναμία είναι οι αγορές και ο πόλεμος μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων. Ε, οι Κινέζοι ε, δεν αγοράζουν πια δολάρια, πουλάνε. Η φορολογική κατάσταση των ΗΠΑ, η δημοσιονομική κατάσταση είναι χειρότερη στις ΗΠΑ από ό,τι στην Ευρώπη. Ε, το ομοσπονδιακό χρέος προστίθεται στο χρέος των, πολιτών, των πολιτιών. το ευρώ είναι φάρος σταθερότητας όπως είπε ο κύριος Τρισέ και θα επιζήσει του κυρίου Βαν Ρόμποϊ διότι η Ένωση είναι η πιο σημαντική οικονομική ενότητα στον κόσμο παρά τα πραγματικά προβλήματα στα οποία αντιμετωπίζει διστακτικά η Ευρώπη. Οι 27 όμως είναι η μεγαλύτερη εξαγωγής και εισαγωγής προϊόντων στον κόσμο. Εξαγωγή, η μεγαλύτερη εξαγωγής υπηρεσιών. Έχουμε την πιο υγιή αγορά. Η Ένωση είναι ο πρώτος προορισμός για τις επενδύσεις τρίτων χωρών. Οι επιχειρήσεις των ε, της Ένωσης έχουν τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επενδύσεις. 5% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει η Ένωση παράγει 30% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η Ιαπωνία 7%, η 25%. Δίνουμε 55% βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες Παρακαλώ να τελειώσετε, ε, λέει η πρόεδρος. Ναι, τελειώνω κυρία μου. Πρέπει να επιβάλλουμε διαφάνεια στα, ε, ε, στις αγορές, διεθνώς για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Ευχαριστώ, ο χρόνος έχει τελειώσει. Κυρία Φέλτ για δύο λεπτά παρακαλώ. Yes, thank you, Chair. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως υπογράμμισε ο συνάδελφος Γκοζές, ορισμένοι μισούν το ευρώ το βλέπουν σαν τη βάση, τη ρίζα του κακού και χαίρονται για να, κατα... να καταρρεύσει η Ευρωζώνη. Αλλά κάνουν λάθος αυτοί. Ζουν στο παρελθόν. Ε, τα σημερινά προβλήματα δεν οφείλονται στο ευρώ. Αντίθετα, το ευρώ μας προστατεύει από τα χειρότερα. Χρειαζόμαστε το κοινό νόμισμα, αλλά χρειαζόμαστε και σωστή διακυβέρνηση της Ευρωζώνης ε, η χαλαρή συνεργασία δεν είναι πλέον επιλογή. Είμαστε σε ένα πλοίο με, μια, με μια τεράστια τρύπα. Ή θα κολυμπήσουμε ή θα βυθιστούμε. Οι εθνικέ κυβερνήσει όμω εξακολουθούν να, μοιάζουν, να θεωρούν ότι φτάνει να φτιάχνουν ομάδε εργασίε, να μιλάνε ίσω στενότερη συνεργασία, αλλά ίσω και όχι κτλ. Τα καλά νέα είναι όμω ότι ενεργούν πιο αποφασιστικά στην περίπτωση της Ιρλανδίας Γερμανίας γιατί χρειάζεται ταχύτατη αντίδραση και είναι ευπρόσδεκτη αυτή. Δεν πρόκειται για τη διάθεση μιας χώρας, πρόκειται για την αξιοπιστία της Ευρωζώνης πρόκειται ε, για μια δοκιμασία, ένα τεστ μας επιβάλλει ο κόσμος αν είμαστε σε θέση να ενεργήσουμε διότι η εμπιστοσύνη του κόσμου στην Ευρωζώνη είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα του νομίσματός μας. Είναι, έτσι μπαίνουν τα λεφτά στην τσέπη μας, δηλαδή από την εμπιστοσύνη που έχουν οι άλλοι. Γι' αυτό παρατρύνω τους εθνικούς ηγέτες να σταματήσουν τα λαϊκίστικα ε, και να μην σκίζουν ευρωνομίσματα δημόσια αλλά να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το κοινό μας νόμισμα. Όσον αφορά τα μέτρα λιτότητας, επικρίνονται πολλοί και ορισμένοι λένε ότι θα ζημιώσει η οικονομία. Βεβαίως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, είναι απαραίτητα όμως τα μέτρα αυτά για να εξηγηθούν τα δημόσια οικονομικά και είναι και ένα σημάδι αλληλεγγύης μεταξύ κρατών της Ευρωζώνης. Δεν πρέπει όμως να μιλάμε μόνο για τις δαπάνες αλλά και για τα έσοδα διότι και εκεί απαιτούνται μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να είχαν γίνει από καιρό. Ευχαριστώ πολύ, ο χρόνος έχει τελειώσει. Ο κύριος Φαντάλεν για ένα λεπτό. Από την εισαγωγή του ευρώ, κυρία Πρόεδρε, η ΕΚΤ δεν είχε περάσει από μια χρονιές τόσο αναστατωμένες ας πούμε όπως αυτή του 2009 πολλές ε, μεγάλος αγώνας αλλά θα πρέπει να αγωνιστούμε ακόμα περισσότερο κατά της κρίσης να, δημιουργούμε, να δημιουργήσουμε ένα πήγον ταμείο εντάξει αλλά ε, τα χρέη συνεχίζονται και δεν επιστρέφονται από χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία Χρειαζόμαστε δημοσιονομική πειθαρχία, μείωση των δαπανών και κυρώσεις. Κυρώσεις λοιπόν. Ο κύριος Μπάλτς ήταν πολύ σαφής από αυτή την πλευρά. Θα ήθελα και το Συμβούλιο λοιπόν να υιοθετήσει το πακέτο ανάπτυξης και σταθερότητας. Τα περισσότερα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου θα θέλανε επίσης αυτά να ισχύσουν και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ε, 2,95% ε, αύξηση είναι γενναιόδωρο. Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί το Ευρωκοινοβούλιο θέλει κι άλλα. Ο κύριος Πάσχα τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία ε, Ο κύριος, κύριε Τρισέ, σύμφωνα με μια αναφορά στο Reuters, φαίνεται ότι είπατε το Σεπτέμβριο ότι αν γνωρίζετε ότι η Σλοβακία δεν θα υποστήριζε την διάσωση της Ελλάδας, δεν θα αφήνατε τη Σλοβακία να μπει στην Ευρωζώνη. Αν ξέρατε ότι θα είχε μια τέτοια αντίρρηση η Σλοβακία. Το γεγονός είναι ότι η Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να πληρώσει, να εξοφλήσει τα χρέη της. Η διάσωση λοιπόν της Ελλάδας πρέπει να είναι προαιρετική υπόθεση, όποιος θέλει. Ε, οι μηνιαίες σας αποδοχές κύριε Τρισέ μπορούν να ταΐσουν εκατοντάδες οικογένειες στη Σλοβακία για ένα μήνα. Δοθέντος αυτού αναρωτιέμαι γιατί νομίζετε ότι πρέπει να εξασφαλίσετε οι φίλοι σας στις τράπεζες και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μπορούν να τρώνε περισσότερο χαβιάρι αφαιρώντας εισόδημα από τους, ε, από τους κατοικούς της χώρας μου. Ο κύριος Φεραρά έχει δύο λεπτά. Η κυρία Φεραρά, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να είχε προχωρήσει με μια κοινή λύση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, κυρίως τις μεγάλες. Και αυτό μάλιστα πριν να ασχοληθεί με άλλες υποθέσεις. Ουσιαστικά σήμερα συζητήσαμε ανοιχτά την πτώχευση κρατών, αλλά δεν έχουμε σαφείς λύσεις ε, για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η ε, παρέμβαση στην Ελλάδα και οι εξελίξεις εκεί καταδεικνύουν ότι η Ευρώπη χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση και η ε, λύση που βρέθηκε είναι μια διμερής λύση που τελικά υπάγει κάθε κράτος σε κρίση από τους ομότιμους, χωρίς αντικειμενικά όμως κριτήρια. Το ΕΚΤ, η ΕΚΤ θα πρέπει να είναι η Άγκυρα. Η Άγκυρα που βοηθάει ε, να μειωθεί η πτυτικότητα ε, στα κρατικά χρέη. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμα. Έχω τρεις ερωτήσεις λοιπόν κύριε Τρισέ. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η θέση της ΕΚΤ σε σχέση με τη σταθερότητα γιατί και σε σχέση με τη δημιουργία πραγματικού αλληλέγγυου μηχανισμού ως προς το δημόσιο χρέος. Δεύτερον, ποιες είναι οι διαφορές που οδήγησαν την ΕΚΤ να μην προσυπογράψει το σύνολο των συστάσεων της Task Force του κ. Βαν Ρόμποϊ. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή ε, Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί να επιβιώσει με παρά τις διαφορές της αναπτυξιακές μεταξύ κρατών μελών χωρίς να έχει κοινό μηχανισμό ώστε να έχουμε συγκερασμό προσπαθειών σας ευχαριστώ και τώρα φτάνουμε στο Catch the Eye. Ο κύριος Κέλλη πρώτα απ' όλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ως Ιρλανδός θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη περηφάνεια για το όσα ακούω σήμερα και είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες μας θέλουν να γίνει ό,τι χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Καταρχά, ευχαριστώ για την υποστήριξη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του Σωματικού Ταμείου, βράχη πρόθεσμα. Δεύτερον και πιο σημαντικό, η αρχιτεκτονική τη εποπτεία των αρχών της Ευρώπης θα πρέπει να λειτουργήσει κατά τρόπο αποτελεσματικό έτσι η σχέση αιτιότητας μεταξύ των ε, τραπεζών που δεν κάνουν στα δουλειά τους, των κυβερνήσεων που δεν είναι αρκετά σταθερές ή αρκετά, ε, δεν έχουν αρκετά σταθερή πολιτική σε ορισμένα θέματα να αντιμετωπιστεί μια διαπαντός. Και πιστεύω ότι με τον τρόπο που στέκεται στο πλευρό μας η Ευρωπαϊκή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να αποτρέψει το χειρότερο. Πολλά μπορούν να γίνουν, πιστεύω, και χρειάζεται βελτίωση σε όλα αυτά τα συστήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κύριε Ντερόσα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε κύριε Πίτρο Περέν και κύριε Τεσέ, μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σήμερα. Μα δώσετε περισσότερε πληροφορίε από ό,τι η Ιρλανδική κυβέρνηση, κύριε Ρεν και κύριε Τρισέ. Η κυβέρνηση μα έλεγε ψέματα επί σειρά μηνών. Ανησυχούσαν περισσότερο με την προάσπιση του ιστορικού του παρελθόντο και τη κληρονομιά του παρά το μέλλον των, και το βιοποριστικό μέλλον των πολιτών τη Ιρλανδία. Εγώ θα ήθελα να εξασφαλίσετε το χρονικό πλαίσιο για την βοήθεια και οι στόχοι για τα χρέη να είναι τέτοιοι ώστε να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικέ πτυχέ για την Ευρώπη και ανάγκη να εξασφαλίζεται ότι η Ιρλανδία να μπορεί να αναπτυχθεί οικονομικά και να δημιουργεί θέσει απασχόληση δεν θα υπονομευτούν. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε επίση ότι κατανοείτε πλήρω ότι η αύξηση του 12,5% του φόρου κερδών επιχειρήσεων τη Ιρλανδία δεν είναι μια λύση για την κρίση τη Ιρλανδία ούτε τη Ευρώπη αλλά θα μπορούσε μάλιστα να δημιουργήσει, να, οικονομήσει, να δημιουργήσει μια έρημο στον αφορά τη απασχόλησης και την οικονομία. Όλοι Σμιτ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Τρισέ και τον κύριο Ρεν για την έξοχη δουλειά που έκαναν αυτού του δύσκολου καιρού που περνάμε. Έχω δύο ερωτήσει, κάποιε ερωτήσει μα συγκεκριμένε. Η χώρα μου δεν ανήκει στην Ευρωζώνη και ακούμε συζητήσεις όπως αυτές που διεξάγονται εδώ σήμερα. Γι' αυτό είχαμε ψηφίσει όχι εμείς στο ευρώ, γιατί είχαμε αμφιβολίες. Και βλέπετε ότι τελικά είχαμε δίκιο. Το ευρώ δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό λέγεται και ακούγεται. Λοιπόν κύριε, έχω μια ερώτηση. Είναι σφαλμένη δήλωση αυτή που ακούω για το ευρώ ή έχει κάποια βάση. Και γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο όσον αφορά το ευρώ, διότι το ευρωπαϊκό αυτό νόμισμα η Ευρωζώνη μπήκαν στο μάτι τη θύελα ή φταίνει οι εθνικέ πολιτικέ στην Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιρλανδία που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Λάθο πολιτικέ που δεν πέτυχαν. Ευχαριστώ, Τζο Higgins, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, σαν Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί εσείς και η, Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδοθήκατε στους κερδοσκόπους και στους καρχαρίες των διεθνών χρηματαγορών, τους επιτρέψατε να δημιουργήσουν πανικό στις αγορές όσον αφορά την αλληλική κρίση, πανικό για να παρέμβετε εσείς, για να δώσετε εγγύησεις και να δώσετε ε, διάφορα δισεκατομμύρια τα οποία αυτοί στοιχημάτισαν σε ε, κακά χρέη. Η Πορτογαλία και η Ισπανία θα είναι η επόμενη. Βάζω στοίχημα. Εσεί και ο κύριο Ρεν παραδοθήκατε στη δικτατορία τη αγορά που είναι ε, ανεξέλεγκτη και ανώνυμη. Το, πόσο το δικαιολογείτε αυτή. Οι ιδιώτε, οι κερδοσκόποι και οι μέτοχοι έπαιξαν δισεκατομμύρια σε ιδιωτικέ συμφωνίε με διάφορου τραπεζίτε στην Ιρλανδία για ιδιωτικά κέρδη. Και όταν απέτυχε το στοίχημα, εσείς υποστηρίζετε την ε, άχρηστη κυβέρνηση της Ιρλανδίας να φορτωθεί στους στοχούς και στους συνταξιούχους που πρέπει να πληρώσουν το κόστος του στοιχήματος και του παιχνιδιού. Και στέλνετε και το Εθνές Νομισματικό Ταμείο σαν στατιώτες του νεοφιλελευθερικού καπιταλισμού για να πληρώσουν η Ιρλανδία. Ηθικά και διαφορετικά δεν πρέπει να πληρώσουν και θα πρέπει να αντισταθούν σε αυτή την καταστροφική επίθεση κατά το, το επίπεδο διαβίωσης και της Δημοκρατίας Ιρλανδίας. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Μπάτμιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Οι εκλογές μου στο Λονδίνο δεν μπορούν να ανεχθούν τις 288 λίρες κατά οικογένεια που είναι το μερίδιό τους για τη συνεισφορά για τα 7 δισεκατομμύρια που δίνονται για βοήθεια στην Ιρλανδία. Οι Ιρλανδοί είναι εκείνοι που δημιούργησαν την κακή τους αυτή η μοίρα. Η κυβέρνησή τους δεν χειρίστηκε σωστά την οικονομία και δημιουργήσει αυτή την ακμή όσον αφορά τα δάνεια που ήταν μια φούσκα. Αλλά ακόμα χειρότερο μπήκαν στο ευρωπαϊκό νόμισμα. Το πρώτο βήμα για να λυθούν τα προβλήματά του είναι να αποχωρήσουν από το ευρώ. Ανταυτού η Ιρλανδία επέλεξε να υποστεί την οικονομική διακυβέρνηση υπό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο πιο πολλοί αργούν να βγουν από το ευρώ, τόσο χειρότερε θα είναι οι συνέπειε όταν βγουν τελικά. Το ίδιο ισχύει βεβαίω και για την Πορτογαλία, για την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα και σίγουρα και άλλους. Το μόνο λογικό πράγμα που, που έκανε η μακαρίτησα η εργατική κυβέρνηση είναι που κράτησε την Βρετανία εκτός ε, του ευρώ. Και η συμμαχία το καλύτερο που θα είχε να κάνει είναι να μην δίνει και άλλα χρήματα για να σώσει αυτούς που σφατάλησαν τα χρήματα αρχικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακίνες είναι η επόμενη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Μπάτεν καλά τα λέει. Η Ιρλανδική κυβέρνηση έκανε κάκιστη διαχείριση των οικονομικών της χώρας και είναι θλιβερή μέρα για τον Ιρλανδικό λαό που αναφερόμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα υπ' αυτές τις συγκεκριμένες περιστάσεις αλλά η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι μια κατάσταση που αλληλεγγύη. Και ίσω δεν το καταλαβαίνει αυτή τη λέξη ο κ. Μπάτεν, τη λέξη αλληλεγγύη. Και η Ιρλανδία, όπω και η Ιρλανδία χρειάζεται την Αγγλία και η Αγγλία την Ιρλανδία και την οικονομία τη. Είμαστε όλοι δεμένοι μεταξύ μα και μην το λησμονούμε. Να θέσω κάποια ερωτήματα, διότι αυτού του φορτισμένου καιρού χρειαζόμαστε ξεκάθαρο κεφάλι και πληροφορίε. Ε, πού, πού βρίσκονται, τι γίνεται, ε, τι έγινε με τις δοκιμές του στρες τελικά για τις τράπεζες και πώς αντέχουν γιατί φαίνεται ότι έχουν το τεστ για τις αντοχές των τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να απαντήσει ποια είναι η εντολή της και κάποιος αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα στις εναρκτήριες δηλώσεις διότι ξανά υπάρχουν σχέσεις, συσχετισμοί μεταξύ όλων των τραπεζών. Των τραπεζών των γερμανικών, των γαλλικών και άλλων χωρών που επένδυσαν σε Ιλλανδικές τράπεζες που πρέπει να δουν τι έκαναν και γιατί έκαναν αυτό που έκαναν. Και τέλος υπάρχει και πολιτική αστάθεια σήμερα το απόγευμα στην Ιρλανδία. Είναι λυπηρό, αλλά είναι αναγκαίο να γίνουν, να διεξαχθούν γενικές εκλογές. Σα ευχαριστώ. Έχει τελειώσει ο χρόνο σας. Η κυρία Γιάκονσάρη έχει ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ίδρυ ο ιδρυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ρόμπερτ Σούμαν, είπε ότι η Ευρώπη δυναμώνει από τις κρίσεις. Θα έπρεπε λοιπόν σήμερα η Ευρώπη να με πολύ γρήγορα, γιατί μία κρίση πέφτει μετά την άλλη. Βεβαίω είναι μεγάλη πρόκληση για το πολιτικό σύστημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Τα προβλήματα της Ιρλανδίας είναι εν μέρη αποτέλεσμα δύναμων κυβερνήσεων. Όμως, αυτό το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι το φάρμακο να μην είναι χειρότερο από την ασθένεια. Ο πράσινος αντιπρόσωπος αναφέρθηκε στην ταχεία αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων στην Ιρλανδία. Αυτό θα οδηγούσε στο θάνατο της οικονομίας της Ιρλανδίας. Δεν μπορούσαμε ποτέ μετά να ξαναπάρουμε τα χρήματά μας. Πρόεδρε, κύριε Τρισέ, γνωρίζουμε όλοι ότι κύριο καθήκον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η διαφύλαξη της νομισματικής σταθερότητας. Το στόχο αυτό μπορείτε να το πετύχετε με τον καλύτερο τρόπο εάν έχετε πολιτική ανεξαρτησία. Και σε αυτό το σας έχουμε υποστηρίζει. Τα τελευταία όμως χρόνια και με τη μεγάλη κρίση α, αναλάβατε και ένα άλλο μεγάλο καθήκον, τη διαφύλαξη σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των χρηματοπιστωτικών αγορών. Και μας και είδαμε ότι αναλάβατε αυτό το καθήκον και το έργο με πολύ μεγάλη ευθύνη, υπευθυνότητα, επαγγελματικό τρόπο. Όμως ε, συνεργαστήκατε αποκλειστικά με κυβερνήσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είχατε απόλυτη πολιτική ανεξαρτησία. Ήσασταν υποχρεωμένοι να ε, ενταχθείτε στη διελκυστήρδα την πολιτική ε, με τις ε, κυβερνήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς σκοπεύετε να διαμορφώσετε, να ζητήσετε μια διαμόρφωση ενός συστήματος διαφορετικού έτσι ώστε να διαφυλάξετε την πολιτική σας ανεξαρτησία. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ε, ομιλήτρια, κυρία Φιγκερίδου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οι ανισορροπίες ενισχύονται, οι διαφορές επιτείνονται μεταξύ των οικονομιών της Ευρωζώνης παρά τις υποσχέσεις, παρά τις προτάσεις. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι το εξής. Δεν πιστεύετε ότι είναι εύθετος πια ο χρόνος να αναθεωρήσουμε τις πολιτικές. Νομίζω ότι επιμένετε με με κράτη που έχουν αδύναμη οικονομία να τηρούν του όρους του Συμφώνου Σταθερότητας και αυτό προκαλεί μεγαλύτερες ασυμμετρίες στην ανάπτυξη, στην ανεργία κτλ. Μήπως είναι σκόπιμο ε, να εξετάσετε την κοινωνική βιωσιμότητα. Αυτή τη βδομάδα στην Πορτογαλία ε, οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται και θα κατέβουν σε ομαδική καθολική διαδήλωση. Ε, λόγω της πολιτικής λιτότητας που θα οδηγήσει σε σοβαρή ύφαση. Ε, λοιπόν, δεν νομίζετε ότι είναι πια καιρός να αλλάξετε πολιτική και να δώσετε προτεραιότητα στην κοινωνική στήριξη, ε, στην έκφραση της ελεγγύης αν όχι τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Το μικρόφωνο τώρα παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ μέρους οποίας θα λάβει το λόγο ο Επίτροπος κ. Ολυρέν. Ε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, πριν από οτιδήποτε άλλο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Ε, πολύ σημαντική ήταν. Η κυρία Γιακονσάρη μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύχθηκε πάντα μέσω κρίσεων. Είναι σωστό αυτό ιστορικά. Απολύτω θα έλεγα μάλιστα. Και αυτή τη φορά και πάλι έτσι έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, μέσω των περιστάσεων, αυτού του τύπου των παραστάσεων αναγκαζόμαστε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε όλες τις απειλές εναντίον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτή την εποχή ε, συνεργαζόμαστε για την Ιρλανδία για να εξασφαλίσουμε το μέλλον αυτής της χώρας ταυτόχρονα προσπαθούμε να οικοδομήσουμε πιο μακροπρόθεσμα ένα πραγματικό ευρωπαϊκό αρχιτεκτόνημα το οποίο θα ενισχύσει την οικονομική μας ένωση και ακόμη θα συμπληρώσει αυτή την ένωση με αυτό τον ε, οικονομικό πυλώνα ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η στόχη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. και γι' αυτό πρέπει να ενεργήσουμε σαν πυροσβέστες τρόπον την για να σβήσουμε τη φωτιά στο δάσος. Αυτό αντιμετωπίζουμε σήμερα. Σκόρπιες φωτιές δεξιά και αριστερά. Και γι' αυτό, πυρκαγιές δηλαδή, και γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε κανόνες ε, η Ιρλανδία βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Ξέρετε κυρία Ιακονσάρη ότι λέμε στην Φιλανδία ότι πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που το χρειάζονται όσο είναι ακόμη καιρός. Ε, και σήμερα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε την Ιρλανδία κατά τη διάρκεια αυτής της δυσχερούς περίοδου. Όχι μόνο για να βοηθήσουμε την Ιρλανδία, αλλά για να εξασφαλίσουμε την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή την εποχή να αμφισβητηθούν ε, να αμφισβητηθεί η ανάπτυξή μας, να δημιουργηθούν δηλαδή στοιχεία που να την απειλούν. Η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να μπορεί να αναπτυχθεί με σταθερότητα και πρέπει να εργαστούμε για την απασχόληση. Γι' αυτό μιλάμε. Μιλάμε για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και της απασχόλησης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για αυτή την ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που μπήκε σε βάθος και συμφωνώ με τον κύριο Κοζές ότι πρέπει πράγματι να εξηγήσουμε καλύτερα γιατί πράττουμε αυτά που πράττουμε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να καθησυχάσουμε τους συμπολίτε μας. Πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση. Ε, υπάρχει παραπληροφόρηση και συνεπώς ο καθένας μας πρέπει να παίξει το ρόλο του επικοινωνώντας τα σωστά μηνύματα και το Ευρωκοινοβούλιο και καθένας από εσά σαν εκπρόσωποι του ε, λαών έχετε ρόλο να παίξετε. Η ιδέα δεν είναι εδώ να βρούμε τον αποδιοπομπαίο τράγο ε, η ιδέα είναι να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα που προστάτευσε τους Ευρωπαίους πολίτες από συνέπειες που θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο επιβαρημένες. Μιλάμε για αποοικοδόμηση του ευρωπαϊκού σχεδίου. Αυτό είναι αδιανόητο. Όλα τα κράτη-μέλη θα βρεθούν σε πολύ πιο δύσκολη, θα ήταν σήμερα σε πολύ ε, δυσχερέστερη κατάσταση χωρίς την Ένωση και χωρίς την πανοπλία, την ασπίδα που προσφέρει. Ε, το ευρώ είναι στο κέντρο της Ευρώπης. Δεν είναι τεχνική ρύθμιση, είναι ένα πραγματικό σχέδιο που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε βαθύτερα με την Ένωση. Συνεπώς, είναι θεμελιώδες να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Κυρία Πρόεδρε, καταλήγω λέγοντας ότι η κυρία Γκουλάχ έκανε ένα πολύ σημαντικό σχόλιο όταν μίλησε για τους βασικούς αρχικούς στόχους των ιδρυτών της ΕΟΚ τότε της Ευρωπαϊκής Νομισματικής και Οικονομικής Ένωσης. Ο κύριος Τρισέ μας μίλησε και αυτός. Γι' αυτά και το νομοθετικό πακέτο είναι στα χέρια σας τώρα άλλωστε και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική, πραγματικά ισχυρή οικονομική ένωση. Έχει οριμάσει ο χρόνος για να συμπληρώσουμε τα κετά και ακριβώς αυτό είναι ο στόχος του νομοθετικού πακέτου ενισχύοντας την διακυβέρνηση και τη διαφάνεια. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δεν υπάρχει πια δυνατότητα να μιλήσετε κάνοντα χρήση τη ε, γαλάζια κάρτα σα. Δεν το επιτρέπει ο κανονισμό. Συνεχίζουμε τη συζήτηση τώρα, όπω το προβλέπει η ημερήσια διάταξη. Κύριο Ρώσα, Ντερόσα, χωρί μικρόφωνο δεν υπάρχει δυνατότητα να παρέμβετε χρησιμοποιώντας τη γαλάζια κάρτα σας σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε κανονισμούς, συγκεκριμένους κανόνες του Κοινοβούλου που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κύριε Τρισό, το λόγο. Uh, Point of order. Διαδικαστικό παρακαλώ. Ένα διαδικαστικό κυρία Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε ε, ε, πρόκειται να συναντηθώ με τους Ιρλανδούς σε σχέση με τα θέματα της χώρας. Αλλά όσο και δύσκολη και αν είναι η κατάσταση στην Ιρλανδία, η συζήτηση εδώ σήμερα είναι για την έκθεση την ετήσια της ΕΚΤ Πολλές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκαν στην Ιρλανδία. Δεν ήταν δυνατόν να απαντηθούν. Ευχαρίστως να συναντηθώ με τους ευρωβουλευτές της Ιρλανδίας για να το συζητήσουμε με λεπτομέρεια αν θέλετε, αλλά όχι εδώ σε σχέση με αυτή την έκθεση. Έχετε το λόγο κύριε, κύριε Τρισέ. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να πω ότι οι ερωτήσεις που τέθηκαν είναι πραγματικά πολύ επίκαιρες και καλύπτουν το σύνολο των θεμάτων, θα έλεγα, που έχουν εξέχουσα σπουδαιότητα σήμερα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ταυτόχρονα σε περισσότερους βουλευτές διότι ε, υπήρχε, υπήρξαν συγκλίνουσες ερωτήσεις. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε υπεύθυνοι για το M του EMU, το M, το monetary, το νομισματικό. Έχουμε συναισθήματα βεβαίως και για το ε, το οικονομικό. Και οι οδηγίες που μας έχουν δοθεί από τους λαούς της Ευρώπης, από το κοινοβούλιο που ψηφίσανε το Μάστριχτ, ε, είναι η σταθερότητα. Πρέπει να δώσουμε σταθερότητα τιμών σε 300 τόσα εκατομμύρια κατοίκους. Όπως εξήγησα λοιπόν πριν από λίγο, τα καταφέραμε να εξασφαλίσουμε σταθερότητα τιμών ακολουθώντας τον ορισμό που είναι ουσιαστικά ο καλύτερος στον κόσμο. Τι είναι ο, ορισμός αυτός, είναι το παγκόσμιο benchmark. Μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε λοιπόν σταθερότητα τιμών στα 12 χρόνια του ευρώ και είμαστε αξιόπιστοι και για τα επόμενα 10 χρόνια σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουμε. Σας το λέω όσο πιο καθαρά μπορώ γιατί πολλές ερωτήσεις που μου απευθύνονται είναι ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την οικονομική ένωση που είναι κομμάτι του EMU αλλά δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την οικονομική ένωση. Έχουμε ιδέες, έχουμε συστάσεις, έχουμε κάποια διαγνωστικά εργαλεία, ε, έχουμε κάνει ανάλυση, αλλά ως εκεί. Δεύτερο σημαντικό σχόλιο. Αντιμετωπίζουμε τη χειρότερη κρίση από το δεύτερο παγκόσμιο ε, πόλεμο παγκόσμια. Αν δεν είχαμε αντιδράσει γρήγορα και θαραλέα, ε, οι κεντρικές τράπεζες και η ΕΚΤ και οι κυβερνήσεις θα είχαμε αντιμετωπίσει τη χειρότερη κρίση όχι από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από, το, από το πρώτο παγκόσμιο ε, πόλεμο γιατί θα είχαμε περάσει σε μεγάλη ύφεση σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάω πρέπει να πω ότι οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια χρειάστηκαν να ενεργήσουν ευρύτατα και ο φορολογούμενος έχει κινητοποιηθεί για να αποφύγει την δραματική ύφεση και αν θέλετε και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού η επιβάρυνση είναι η ίδια δεν χρησιμοποιείται για δαπάνες αλλά για ζημίες. Εν πάση περιπτώσει πρόκειται για τεράστια προσπάθεια. Αλλιώς θα ήταν δραματική η κρίση. Αυτό βεβαίω σημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομία και η χρηματοπιστωτική αγορά είναι πάρα πολύ εύθραυστη και πρέπει να βρούμε τρόπους να ρυθμίσουμε αυτό το εύθραστο πλέον. Αλλά δεν είναι ευρωπαϊκή κρίση. Είναι η επιπτώσεις στην Ευρώπη. Οι επιπτώσεις από μια παγκόσμια κρίση. Και ε, το ίδιο μπορεί κανείς ε, να σκέφτεται τι να κάνει δηλαδή στη ΣΥΠΑ ή στην Ιαπωνία. Ε? Μιλάμε για τις δύο άλλες πολύ προχωρημένες οικονομίες. Έχουν και αυτοί τεραστίου μεγέθους προβλήματα. Πρώτου μεγέθους αν όχι τεραστίου. Λοιπόν, να μην μετατρέπουμε την νόμιμη ανάλυση του πώς να τρέξουμε επιτυχημένα την οικονομία και να τη μετατρέψουμε σε επίκριση του ευρώ που το ευρώ απέδωσε ακριβώς αυτό που αναμενόταν όπως σας είπα. Θα ήθελα ακόμη να πω ότι όταν εξετάζω την υποσυνομική κατάσταση των πιο προχωρημένων οικονομιών Μπορώ να πω ότι η Ευρώπη και η Ευρωζώνη ειδικότερα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι η Ιαπωνία και είπα όσον αφορά την χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους γύρω στο 6% ίσως λίγο λιγότερο ε, συγκεντρωτική φορολογική θέση δηλαδή Δέκα ή περισσότερο είναι το ποσοστό στις δύο άλλες ε, προηγμένες χώρες. Σας δίνω τις διαστάσεις των μεγεθών δηλαδή. Έχουμε λοιπόν τι κακή συμπεριφορά από διάφορες χώρες που δημιουργούν προβλήματα μέσα στη χώρα τους βεβαίως αλλά από τα οποία προβλήματα προκύπτει χρηματοπιστωτική αστάθεια. Δεν είναι το ευρώ που περνάει την κρίση είναι η χρηματοπιστωτική αστάθεια που έχει προκύψει από την κακή συμπεριφορά μέσω φορολογικής πολιτικής. Και έχουμε την αλληλοεπίδραση των αγορών βεβαίως. Είμαστε οικονομίες των αγορών. Βασικά λοιπόν η διάγνωσή μας είναι ότι αυτό που είναι αφύσικο στη λειτουργία της Ευρώπης ήταν η κακή οικονομική διακυβέρνηση των, της Οικονομικής Ένωσης. Και με θλίψη μου λέγω ότι αυτό δεν με εκπλήσει. Διότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης επεκρίθη εσφαλμένα από κάποιους από την αρχή. Και θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι εγώ ίδιος ενημέρωνα το κοινοφούλιο για τη μάχη που δίναμε, διότι μεγάλες χώρες ήθελαν να διαλύσουν το σύμφωνο αυτό ή να το αποδυναμώσουν πολύ. Και δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι ήταν οι μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης που το ήθελαν αυτό και ότι οι μεσές και οι μικρές χώρες αντιστεκόταν σε αυτή την τάση. Το 2004 και το 2005 συνέβη αυτό. Θα θυμόσαστε ότι έγινε σκληρή μάχη. Διότι πήγαμε στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και από τι φόρο τιμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ήταν υφάλια τότε, πιο υφάλια από το Συμβούλιο και υποστηρίζαμε εμεί πλήρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έπρεπε να το θυμίσω σε όλου μα αυτό. Άκουσα διάφορε ερωτήσει σχετικά με το τι ζητούμε σε αυτή τη φάση και τι στόχο έχουμε. Είχαμε ήδη πει όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τι προτάσει τη ότι θεωρούσαμε ότι δεν αρκούσαν οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπόψη αυτό που αισθανόμαστε, αυτό που βλέπουμε όσον αφορά τη λειτουργία της Ευρώπης εν γέννη και των 27 συν τις 16-17 ε, χώρες της Ευρωζώνης θα έλεγα ότι η πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ αδύναμη όσον αφορά τον αυτόματο χαρακτήρα των μέτρων και την αυστηρότητα της διακυβέρνησης και όσον αφορά την εποπτεία στο φορολογικό τομέα και όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα ε, όσον αφορά την εποπτεία και τις ανισορροπίες. Και η παρούσα κατάσταση, η παρούσα πρόταση που κάνει το Συμβούλιο στις παρούσες συνθήκες αποδυναμώνει έτσι περαιτέρω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα το μόνο που μπορούμε να πούμε σε εσά αξιότιμοι βουλευτές είναι ότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις περιστάσεις. Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρή εποπτεία πολύ στεναρή διακυβέρνηση. Το 2005 εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου είχα πει ότι δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από την τότε θέση του Συμβουλίου και από αυτό που έγινε τελικά δεκτό. Δεν θέλω να πω περισσότερα, διότι θα έχουμε και άλλες επαφές μεταξύ μας και σημείωσα κυρία Γκουλάγ αυτό που είπατε δηλαδή για την πολύ σκληρή δουλειά που κάνει το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να καταλήξουμε τελικά στη θέση που θα έχει η Ευρώπη. Είναι σαφέστατο το μήνυμά μας όσον αφορά αυτό το θέμα. Για ένα λεπτό να στραφώ στην ανακοίνωση και επικοινωνία μάλλον. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις επικοινωνίες, την επικοινωνία, αλλά όσον αφορά τη δική μας θέση δίνουμε σαφή ορισμό της σταθερότητας τιμών που επιτρέπει σε όλους να κρίνουν τι κάνουμε πάντα τι κάνουμε σε πραγματικό χρόνο. Θα ήθελα να πω ότι ήμασταν η πρώτη, η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που ε, καθιέρωσε αμέσως μετά το Διοικητικό Συμβούλιο συνεντεύξεις τύπου. Και δίνουμε μια εισαγωγική δήλωση που κάνει μια διάγνωση της καταστάσεως ε, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο υπεύθυνοι όσον αφορά την επικοινωνία και την ενημέρωση. Το μόνο που δεν κάνουμε είναι να δημοσιεύουμε τις διάφορες ξεχωριστές θέσεις των διαφόρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικότατο ο φορέας που ε, ε, το νόμισμα αυτό για τα 16 κράτη που είναι κυρίαρχα κράτη αλλά ενωμένα εντός Ευρώπης ότι είναι καλύτερο το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του, σαν σύνολο, ενιαίο σύνολο να φαίνεται ότι είναι ο φορέας, ο αρμόδιος που παίρνει τις αποφάσεις. Ε, ακούστηκαν αρκετές σημαντικές, πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Να πω κάτι σχετικά με το σχόλιο που έλεγε ότι είμαστε υπεύθυνοι για την οικονομία είναι τα κράτη-μέλη. Εμεί είμαστε υπεύθυνοι για το νόμισμα. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη την οικονομία όπως το κάνει κάθε ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα. Αν η οικονομική πολιτική και η φορολογική πολιτική είναι ορθή και λογική, η νομισματική πολιτική που οδηγεί σταθερότητα των τιμών είναι ευκίνητη. Αν θέλουμε κακή οικονομική πολιτική, τότε επιβαρύνεται υπερβολικά ο τομέας ο νομισματικός και αποφάσει πρέπει να πάρει η Κεντρική Τράπεζα. Θα μπορούσα να πω το ίδιο όσον αφορά την διαδραστική επαφή που υπάρχει με τις ε, ε κυβερνήσεις. Υπάρχει σταθερή όμως σχέση. Έπρεπε να λάβουμε διάφορα έκτακτα μέτρα. Και όπως εξήγησα, το κάναμε αυτό για να διαβιβάσουμε, να μεταβιβάσουμε τους παλμούς της νομισματικής μας πολιτικής όπως γινόταν σε αυτές τις περιστάσεις όταν οι αγορές δεν λειτουργούσαν εύρυθμα. Και γι' αυτό οι αποφάσεις που λαμβάναμε όσον αφορά τα επιτόκια δεν διαβιβιζόταν σωστά στην οικονομία, δεν είχαν τη σωστή επιρροή στην οικονομία. Αυτή είναι η ουσία των εκτάκτων μέτρων, των μη τυπικών μέτρων. Βοηθούν στην αποκατάσταση πιο κανονικής λειτουργίας της, νομιζ... διαβίβασης των διάβλων διαβίβασης της νομισματικής πολιτικής. Το ξεκαθάρισα αυτό, το επανέλαβα και σε κάποιο συμπόσιο που εδιεξήχθη. Το καταστήσαμε σαφέστατο. Ποια είναι η διάκριση μεταξύ των κανονικών, των συνηθισμένων μέτρων που αφορούν τη νομισματική πολιτική και των εκτάκτων μέτρων, των εκτάκτων μέτρων που προσπαθούν να βελτιώσουν τη διαβίβαση και την επιρροή που έχουν τα νομισματικά μέτρα. Σημαντικό ερώτημα επίσης ετέθη από τον κύριο Γκοζές όσον αφορά την επικοινωνία και την κοινοποίηση και την, ε, που ανέφεραν κι άλλοι. Υπάρχει μια τάση σε κάποιους διάβλους επικοινωνιών να θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι αποδιοπομπέως τράγος. Αν όλα πάνε κακά, φταίει η Ευρώπη. Ξέρουμε ότι είναι ασφαλμένο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το γνωρίζει προφανώ καλύτερα από όλου του άλλου. Υπάρχει και μια τάση να λέγεται ότι αν όλα δεν πάνε καλά φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φταίει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακόμα καλύτερα φταίει το ευρώ. Αυτό είναι κλασικό φαινόμενο του αποδιοπομπέου τράγου. Το ευρώ σαν νόμισμα είναι το νόμισμα που διατήρησε τη σταθερότητά του εσωτερικά και εξωτερικά με αξιοσημείωτο τρόπο. Δεν είπα εγώ ότι ήταν πιο αξιοσημείωτο από αυτό που έγινε εντός των ιδρυτικών χωρών της, ε, του ευρώ. Καμία κεντρική τράπεζα ε, τα 50 τελευταία χρόνια δεν, έκανε, δεν έλαβε τέτοια μέτρα. Βλέπουμε λοιπόν ένα νόμισμα το οποίο είναι στέρεο στέρεο ε, και σε ιστορικό επίπεδο. Και θα πρέπει να διαφυλαχτούμε, να προφυλαχτούμε από το φαινόμενο δύο πομπέου τράγου. Και θα πρέπει όλοι να εργαστούμε γι' αυτό. Είμαστε, έχουμε πολλή δουλειά όσον αφορά την επικοινωνία και την εικόνα. Λαμβάνω το μήνυμα που αφορά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα και όλες, δηλαδή όλες τις κεντρικές τράπεζες που ανήκουν στην Ευρωζώνη. Είναι ένα πρόβλημα που τίθεται και σε επίπεδο 27 για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ε, λεπτομερή ε, απάντηση την οποία ε, κάνατε αλλά υπό αυτά σε συνθήκας ήταν σκόπιμο να υπάρχει μία λεπτομερής παρουσίαση και τώρα έχει το λόγο ο για δύο λεφτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, και εγώ όσον αφορά τον κύριο Τρισέ, τον Επίτροπο Ρεν και τους συναδέλφους ευχαριστώ όλους για αυτή την ε, συζήτηση η οποία ήταν πολύ αντικειμενική παρόλο που ε, επεκράτησαν και συγκινήσεις των Ιρλανδών συναδέλφων μας αλλά τους καταλαβαίνω. Καταρχήν όσον αφορά την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Κεντρικής Τράπεζας. Ήταν καλό ότι ο Χέλμουτ Κόλ ε, επέβαλε την, ε, ε, την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διότι η τράπεζα αυτή μπόρεσε να στηρίξει να έχουμε μια σταθερή κατάσταση ιδίως τους τελευταίους μένους. Γι' αυτό και πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη και τους επόμενους μήνες για να μπορέσουμε μπορέσουμε να προχωρήσουμε διότι τελικώς εσείς σαν πρόεδρος ε, θα πρέπει να είστε εγγυητής αυτής της ανεξαρτησίας. Επίσης όσον αφορά τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να τους εξηγήσουμε καλύτερα πώς έχει κατάσταση και αυτές οι εξηγήσει δεν πρέπει να γίνονται στην ξύλινη γλώσσα των Βρυξελών αλλά θα πρέπει ε, να εφόσον απευθυνόμαστε απευθυνόμαστε στον απλό άνθρωπο να μιλάμε και ανάλογα. Αναφερθήκατε επίσης στη Βασιλεία 3 κύριε Πρόεδρε και από αυτού μπορώ να τονίσω ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε σύντομα την ε, Βασιλεία 3 αλλά αυτό θα μπορέσει να γίνει μόνο εάν όλοι ε, συνεργαστούμε. Δεν μπορεί εδώ να προχωράει η Ευρώπη μόνη της και εμείς ε, να βασιζόμαστε στην ανταγωνιστικότητά μας. Δηλαδή ε, θα πρέπει ε, η Ευρώπη είτε να εφαρμόζει τα συμμεφωνημένα αλλά εν πάση περιπτώσει διαφορετικά να ε, επιζητήσει άλλες λύσεις. Ευχαριστώ. Έληξε η συζήτηση και το αύριο θα γίνει η ψηφοφορία.